Εκθέσεις της κυρίας Ελισάβετ Βόζενμπεργκ στα δεδρομία των γυναικών στις επιστήμες και τα πανεπιστήμια. Καταρχάς. Και παρακαλώ την κυρία Βόζενμπεργκ να λάβει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, με ιδιαίτερη χαρά θα παρουσιάσω για τελευταία φορά την έκθεσή μου που αναφέρεται στα εμπόδια που ορθώνονται στις φιλοδοξίες των γυναικών να κατακτήσουν τα ανώτατα αξιώματα στην έρευνα την τεχνολογία στην επιστήμη στα διοικητικά συμβούλια σε θέσεις ευθύνης και είναι η τελευταία φορά που μοιράζομαι κάποιες σκέψεις μαζί σας ελπίζοντας τη στήριξή σας αύριο στην ψηφοφορία αυτής της εξαιρετικά προκλητικής και φιλόδοξης έκθεσης ως προς το αντικείμενο όταν μιλάμε για εμπόδια τα οποία χαρακτηρίζονται ονομάζονται ως γυάλινες οροφές ο τίτλος η ονομασία δεν είναι καινούριο, είναι εδώ και 30 χρόνια και θέλει να καταδείξει σε ποιες κατηγορίες εντάσσονται αυτά τα εμπόδια που πραγματικά δεν αναγνωρίζουν τις ίσες ευκαιρίες τις δίκαιες ευκαιρίες που δικαιούνται οι γυναίκες όταν έχουν προσόντα ικανότητες και δεξιότητες να επιδιώκουν φιλόδοξα και έντιμα και ηθικά κάποιου συγκεκριμένους στόχους στα ανώτατα αξιώματα ξεκινώντας θα ήθελα να εστιάσω στους λόγους που γεννήθηκαν αυτά τα εμπόδια και πώς ιδρύονται αυτές οι γυάλινες οροφές όπως λέγονται οι γυάλινοι φραγμοί. οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών οφείλονται αφενός μεν στις προκαταλήψεις που υπάρχουν στην κοινωνία μας και δεν έχουν εξαλειφθεί ακόμη παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο 2015 σε μια κοινωνία εξαιρετικά φιλόδοξη την ευρωπαϊκή που κάθε άλλο παρά την τιμά να έχει τέτοιες διακρίσεις σε βάρος του μισού πληθυσμού του πλανήτη των γυναικών. η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στις οικογενειακές υποχρεώσεις που εκ των πραγμάτων και αυτές ορθώνονται ως εμπόδια όταν αφαιρούν τον χρόνο που απαιτείται από τις γυναίκες αυτές που έχουν τα προσόντα στα οποία προαναφερθήκαμε να επιδιώκουν στόχους έτσι ως αποτέλεσμα βλέπουμε μια ουσιαστική υποεκπροσώπηση στην επιστήμη στην τεχνολογία και ιδιαίτερα σε διοικητικά συμβούλια εκεί όπου οι ηγετικές θέσεις θα πρέπει να επιδιώκουν κάποιες γυναίκες να απαιτούν περισσότερο ανταγωνιστική διάθεση υπό την προϋπόθεση όμως ότι και το περιβάλλον επιτρέπει αυτόν τον ανταγωνισμό να αναπτύσσεται απαριθμώντας κάποια από τα εμπόδια στην επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών τα έχω αριθμίσει σε τέσσερις κατηγορίες τις πιο σημαντικές η μητρότητα εκ των πραγμάτων που από τη φύση είναι προνόμιο και ιδιαίτερο χάρισμα της γυναίκας ορθώνεται ως εμπόδιο όταν απασχολεί τόσο χρόνο στον οποίο θα μπορούσαν οι γυναίκες αυτές η γυναίκα η οποία τιμάται με τη μητρότητα να αφιερώσει στην εξέλιξη των φιλοδοξιών της. αυτό όμως δεν θα έπρεπε να ορθώνεται ως εμπόδιο και ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχουν κάποιες σκέψεις στερεοτύπων του τύπου ότι όταν αφαιρείται ο χρόνος τον οποίο από τη φύση της έχει μια γυναίκα να αφιερώσει στη μητρότητα ε, ε, είναι ε, δυσανάλογος με τον χρόνο που θα έπρεπε να αφιερώσει για να επιδιώξει τους στόχους της η δεύτερη κατηγορία είναι ένα στερεότυπος και εντελώς αναχρονιστικός διαχωρισμός ανάμεσα σε γυναικεία και ανδρικά επαγγέλματα όταν γνωρίζουμε πια ότι όλα αυτά τα κάστρα έχουν κατακτηθεί από τις γυναίκες και μάλιστα με εξαιρετικά σημαντικά αποτελέσματα και επιτεύγματα για την επιστήμη και την τεχνολογία. το μισθολογικό χάσμα που υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναικών που τις οθεί σε πολλές περιπτώσεις να αναφέρονται στα δικαστήρια για να επιδιώξουν την ισότητα και η άνηση πρόσβαση των γυναικών σε συναφή επαγγέλματα στα ερευνητικά προγράμματα. γι' αυτό και οι πρακτικέ που προτείνουμε στην έκθεσή μα αναφέρονται στη μητρότητα στι υποδομέ, στα προγράμματα στη χρηματοδότηση και αναφέρονται βεβαίω και κατατείνουν στι αρχέ και τι αξίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των κρατών μελών που θα πρέπει να υπηρετήσουν το ευρωπαϊκό ινστιτούτο ερευνών και τον ορίζοντα. 2020. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, το βασικότερο όμω οφείλεται, τελειώνω αμέσω, κύριε Πρόεδρε, σε δύο άξονε. Στο προφητόριο που λέγεται οικογένεια και την παιδεία. από εκεί γαλουχείται οι νέοι άνθρωποι της εφηβείας με τις νοοτροπίες εκείνες που θα αναγνωρίζουν ίσες ευκαιρίες στο μισό του πλανήτη με το άλλο μισό του πλανήτη στους άντρες και τις γυναίκες οι οποίοι είναι ανθρώπινα όντα. σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, θα περάσουμε τη διαδικασία Catch the Eye. Αυτή τη φορά θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Κάκια. Grazie, Sir President. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τις ικανότητες ε, όλων ανεξαρτήτως φύλου ε, διασφαλίζοντας τα εξής. Ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, θα λαμβάνουν εκπαίδευση στα ίδια ε, μαθήματα από μικρή ηλικία. Οι εκπαιδευτές από την άλλη μεριά θα πρέπει να τα ενθαρρύνουν να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους ανεξαρτήτως στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Επίσης θα πρέπει να δίνεται περισσότερος επαγγελματικός προσανατολισμός και στα δύο φύλλα τα σχολεία θα πρέπει να βοηθούνται να αγοράζουν το σχολικό υλικό το οποίο είναι απαραίτητο έτσι ώστε τα παιδιά να μάθουν φτιάχνοντας, να μάθουν παράγοντας. Ε, τα κορίτσια θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν θετικές επιστήμες και αυτές που το κάνουν να αποτελούν role models. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Eh, Ο λόγος του κύριο Ρικάρδο Σεραουσάντος. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως ε, καθηγητής και επιστήμονας στην Πορτογαλία έχω δει την αύξηση, σταδική αύξηση του αριθμού των γυναικών στις θετικές επιστήμες και στην επιστήμη. Αυτό ακολουθείται από ότι ακολουθήθηκε από σημαντική βελτίωση του επίπεδου της εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια και στα σχολεία. Παρ' όλα αυτά αναγνωρίζω πως ε, αυτό δεν μπορεί να γενικευθεί ε, και Παρόλο που σε ορισμένα πανεπιστήμια έχουμε ίσο αριθμό γυναικών και ανδρών, αυτό δεν μπορεί να γίνει και σε όλη την κοινωνία, εξαιτία πολλών παραγόντων, όπω για παράδειγμα η μητρότητα και άλλοι. Ε, η εγκυμοσύνη πολύ συχνά δεν μπορεί να συμβιβαστεί με επαγγελματική καριέρα. Θα πρέπει να διευκολύνουμε τις γυναίκες σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό το λόγο χειροκροτώ, επικροτώ και υποστηρίζω αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νότης Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, αφού συγχαρώ την εισηγήτρια, την κυρία Βόζεμπερκ, για την έκθεσή της, θα ήθελα να επισημάνω ότι όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, ακόμη και σήμερα το ποσοστό των γυναικών ερευνητών σε επιχειρήσεις φτάνει το 19%, ενώ παρατηρούνται αντίστοιχα χαμηλά ποσοστά και στον εκπαιδευτικό χώρο είναι εμφανέ ότι τα ποσοστά αυτά προκύπτουν από τις διακρίσεις που γίνονται ει βάρο των γυναικών στους συγκεκριμένους χώρους εργασίας και οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν συχνά σε άνηση μεταχείριση αλλά και σε μισθολογικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα. η διάκριση αυτή αποτελεί παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ω εκ τούτου πρέπει να καταπολεμηθεί συγκεκριμένα θα πρέπει η επιτροπή μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκστρατιών να καταρρύψει όλα τα στερεότυπα που υπάρχουν ει βάρο των γυναικών αλλά και να ενθαρρύνει τι γυναίκε να κατευθυνθούν προ τον επιστημονικό και ακαδημαϊκό χώρο εργασία. τέλος θα πρέπει τα κράτη μέλη μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης να συμβάλλουν στην εξάλληψη των στερεοτύπων που υπάρχουν για τα δύο φύλλα. με αυτές τις προϋποθέσεις θα μπορέσει να μειωθεί το πρόβλημα της διάκριση των δύο φύλων στους χώρους της επιστήμης και της εκπαίδευσης. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Λάουρα Φρέντσα. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι νιώθω ότι με αφορά άμεσα η συγκεκριμένη έκθεση διότι είμαι ερευνήτρια ε, με σύμβαση ορισμένου χρόνου και έχω νιώσει η ίδια το θέμα το οποίο συζητούμε. Η πραγματικότητα είναι δύσκολη στα Ιταλικά πανεπιστήμια, πιο δύσκολη από, τα, ε, από την πραγματικότητα σε άλλες χώρες. Θα ήθελα να σταθώ σε λίγο από τα, αυτά τα στοιχεία για τα όρατα εμπόδια. Ε, στα πανεπιστήμια όλης της Ευρώπης ε, έχουμε όλο ένα και περισσότερο εκδίωξη της ευφυΐας των γυναικών. Στην Ιταλία η πρόνοια και η δυνατότητα να επιλέξουμε και τι θα είναι το αντικείμενο της έρευνάς μας και τι θα είναι το αντικείμενο των σπουδών μας. Θεωρώ ότι πρέπει ταυτόχρονα να καθορίσουμε τι πρέπει να γίνεται στην έρευνα σε πανεπιστημιακό επίπεδο και να υπάρχει και ένα σύστημα πρόνοιας και για τις γυναίκες στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Φρέντσα. Και τώρα η κυρία Λεγκρίπ. Παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τη συνάδελφο ε, την κυρία Βόζεμπερ για την εξαιρετική της έκθεση και για το γεγονός ότι ε, επεσήμανε αυτό το αόρατα εμπόδια, αυτή τη γυάλινη οροφή που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίες ε, γυναίκες στην επιστημονική του σταδιοδρομία. Πιστεύω ότι όλοι μαζί, εάν συνειδητοποιήσουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό, το ανθρώπινο ταλέντο των γυναικών φορές παραγωνίζεται, πολλές φορές ε, αφήνεται στην άκρη ε, και το λάβουμε σοβαρά υπόψη, θα μπορέσουμε να κάνουμε σημαντικές προσπάθειες ώστε να επιτρέψουμε να ε, παρακάμψουμε αυτά τα όρατα εμπόδια και να μπορέσουμε να ε, μην χρησιμοποιούμε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που υπάρχουν παραδοσιακά. Αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει από την ίδια την οικογένεια, από τους γονείς, από τις ίδιες τις κοπέλες, οι οποίες θα πρέπει να μάθουν να ε, ακολουθούν επιστημονικές σταδιοδρομίες και να μην υπάρχουν πλέον αυτά τα στεγανά που υποθέτουν ότι οι άνδρες είναι αυτοί οι οποίοι είναι καλοί στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες και ε, οι γυναίκες μπορούν να δείξουν απλώς ε, εμπάθεια σε κάποιες άλλες επιστήμες. Πρόκειται για στερεότυπα τα οποία θα πρέπει ε, να πάψουν να υπάρχουν και να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες των γυναικών προς όφελος όλων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ έχω ενσυναίσθηση εδώ και Πρόεδρε, δεν κατάλαβα σε ποιον δώσατε το λόγο, γι' αυτό δεν ε, ξεκίνησα. Καταρχά λοιπόν ευχαριστώ την Ελισάβετ Βόζεμπερ και την έκθεσή τη. Αν και δεν μπορώ να υποστηρίξω σε όλα τα σημεία το κείμενο, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με τομεί που ξεπερνούν τι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, σημειώνει πολλά καλά σημεία η έκθεση, ιδιαίτερα στον ε, ακαδημαϊκό και πανεπιστημιακό χώρο. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν οι τροπολογίες μου που ιδιαίτερα δίνουν έμφαση στην επιστήμη και την έρευνα. Εάν μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα των, ε, της διαφοράς αντιμετώπισης μεταξύ των φύλων, θα έρθει η ώρα να συζητήσουμε και το θέμα των οικογενειών και της ανατροφής των παιδιών, όπου βλέπουμε ήδη μια ε, μεροληπτική αντιμετώπιση ως προς την επαγγελματική ή πανεπιστημιακή μόρφωση. Αυτό πρέπει να αλλάξει και για μας εδώ στην Ευρώπη. Η εποχή της ε, μόρφωσης ε, του σχολείου είναι εποχή απόκτησης γνώσεων και πρέπει αυτό να θεωρηθεί όχι μειονέκτημα για τις ε, κυβερνήσεις, κόστος δηλαδή, αλλά κέρδος, όπως άλλωστε και η περίοδος της εξοδότησης. Νομίζω ότι χρειάζεται λοιπόν περισσότερη υποστήριξη για τα παιδιά και για τους γονείς. Ευχαριστώ θερμά. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Γκέρικε. Και τώρα, κύριος Σεβαστιάν. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Όπως λέει η έκθεση, στον ακαδημαϊκό και τον επιστημονικό τομέα δεν πρέπει να θεωρούμε ότι υπάρχει μια εξαίρεση ό,τι αφορά σε σχέση με τους άλλους τομείς της Ευρώπης. Ε, μερικές φορές η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερα γιατί ε, οι γυναίκες που έχουν εκπαιδευτεί επιτυχώ είναι πολλές και περισσότερο από τους άντρε πολλέ φορέ, αλλά δεν αναλαμβάνουν ψηλότερες θέσει. Ε, υπάρχει αυτή η γυάλινη οροφή. Οι τροπολογίες μας που έγιναν δεκτές ε, υπογραμμίζουν ότι για να αποφύγουμε τις διακρίσεις θα πρέπει να λάβουμε μέτρα ιδίως εκπαιδευτικά στα οποία να συμπεριλαμβάνουν και τη συμμετοχή του άντρα σε γυναικείες, θεωρούμενες γυναικείες δουλειές, όπως για παράδειγμα η εκπαίδευση των παιδιών. Αν η γυναίκα αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες της οικογενειακής ζωής, είναι αδύνατο να αποφύγουμε τη γυάλινη οροφή, όσες ποσοστώσεις και αν επιβάλλουμε. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν την συγγήτρια και ελπίζω ότι θα υλοποιηθούν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία προτείνονται. Ευχαριστώ. Now it's time for our guest. On behalf of the European Commission, εκ μέρους της Επιστροπής ε, ο, ο κ. Ναύρασιτς. Speaker, honorable members, first... Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την συγγήτρια την κυρία Βόζεμπερκ από την Επιτροπή Γυναικών για αυτή την πρωτοβουλία. Ε, η έκθεση αυτή για τη σταδιοδρομία των γυναικών σε επιστήμες και στα πανεπιστήμια είναι καλοδεχούμενη. Καταγράφει σωστά την κατάσταση και κάνει πολύ κέρυες προτάσεις. Να σας πω ποιες είναι οι δικές μου σκέψεις. Καταρχήν, θεσμικές ε, ε, αλλαγές. Όπως λέτε πολύ σωστά στην έκθεσή σας, χρειάζονται. Χρειάζεται ε, να καταργήσουμε τους ε, θεσμικούς φραγμούς. Ε, οι γυναίκες μπορεί να έχουν στην επιστήμη τα ίδια προσόντα αλλά δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες επιτυχίες εξαιτίας των στερεοτύπων σε ό,τι αφορά το ρόλο και τις ικανότητές τους καθώς επίσης και εξαιτία των διακρίσεων. Υπάρχουν συμπεριφορές που δημιουργούν τέτοιου είδους προβλήματα. Θεσμικές αλλαγές μπορούν να εξασφαλίσουν ότι ερευνητικά ιδρύματα θα δίνουν ίδιες ευκαιρίες σε άνδρες και γυναίκες σε όλα τα επίπεδα. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ε, στον ευρωπαϊκό ερευνητικό τομέα, τα ερευνητικά ε, όργανα ε, υποχρεώνονται να ακολουθούν μια πολιτική μη διάκρισης και να καταργήσουν τις μεροληψίες, να παρακολουθήσουν την πρόοδο και να έχουν στόχους. Από τα προγράμματα που επικεντρώνονταν σε γυναίκες έχουμε μετακινηθεί ε, διότι δεν ήταν βιώσιμα μακροπρόθεσμα. Ε, οι θεσμικές αλλαγές στα ερευνητικά ιδρύματα αποτελούν το ακρογωνίο λίθο της πολιτικής ισότητας μεταξύ των δύο φύλων στην έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον ορίζοντα 2020 ε, αυτές οι θεσμικές αλλαγές αποτελούν βασικό στόχο. Όμως πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα και καλύτερα θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν την ίδια κατεύθυνση που ακολουθούμε και εμείς. Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας υποστηρίζει. Ο ρόλος σας και η βοήθειά σας είναι χρήσιμα. Δεύτερον, είναι σημαντικό να ενισχυθεί το κανονιστικό πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την ισότητα των δύο φύλων. Λέτε και εσείς στην αρχή της έκθεσής σας ότι... Ε, το λέτε και εσείς στην αρχή της έκθεσής σας και συμφωνούμε. Δεν αρκεί να έχουμε νόμους. Χρειάζεται αυτοί να εφαρμόζονται αποτελεσματικά και να ελέγχεται η εφαρμογή τους. Η Κομισιόν παρακολουθεί την σωστή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη. Στην έρευνα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις, ιδιαιτερότητες, του τομέα, ο οποίος εκτείνεται και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Το Μάιο του 2015 το Συμβούλιο υιοθέτησε τον οδικό χάρτη για τον ε, Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και κάλεσε την Κομισιόν για τα κράτη-μέλη να εφαρμόσει δράσεις προτεραιότητας μέσω προγραμμάτων δράσεων. Η υλοποίηση, ε, η μετατροπή της νομοθεσίας σε πρόγραμμα δράσης είναι πολύ σημαντική. υπάρχουν θέματα τα οποία από τον δικά της εθνικής και της κοινωνικής νομοθεσίας ξέρουμε ότι οι εθνικές στρατηγικές και τα εθνικά κίνητρα δίνουν ε, όθηση στα ερευνητικά ιδρύματα. Τα ερευνητικά ιδρύματα είναι αυτά που τελικά είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των θεσμικών αλλαγών μέσω σχεδίων ισότητας των δύο φύλων. Το Συμβούλιο άσκησε, ζήτησε να παρακολουθείται η πρόοδος μέσω συγκεκριμένων αριθμητικών δικτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί πλήρως. Το εγχειρίδιο για τα βασικά νούμερα του 2015 δημοσιεύτηκε το 2015 ενώ η τελική έκθεση θα δημοσιευθεί τον Ιανουάριο του 2016. Σε αυτή μας την προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να ε, υπογραμμίσει την ανάγκη τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν πλήρως προκειμένου τα στοιχεία που θα μας συλλέξουμε να είναι ε, ε, άψογα. Ε, η ίση συμμετοχή των ανδρών και των γυναικών στα ερευνητικά ιδρύματα είναι πάρα πολύ σημαντική. Η συμμετοχή των γυναικών. Τα, οι γυναίκες αυτή τη στιγμή υποεκπροσωπούνται στην λήψη των αποφάσεων. Και το φαινόμενο αυτό δεν θα διορθωθεί από μόνο του πολλά κράτη-μέλη θέτουν στόχους ή ποσοστώσεις. Το 2013 18 κράτη-μέλη ε, είχαν τέτοιου είδους μέτρα, 8 μόνο το 2008. Χρειάζεται να βελτιώσουμε την ε, ισορροπία των δύο φύλων στην λήψη αποφάσεων. Να σας αναφέρω, να σας αναφέρω τρεις σημαντικές πρωτοβουλίες στην ισότητα των δύο φύλων. Πρώτον, ε, η ισορροπία, ε, η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την, με οικογενειακή ζωή. Έχουμε προετοιμάσει ένα οδικό χάρτη για την βελτίωση αυτής της ισορροπίας ε, και θα ελπίζουμε ότι η αποφάση θα ληφθεί το 2016. περιλαμβάνει νομοθετικά και μη νομοθετικά, νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες. θα ξεκινήσουμε την διαδικασία διαβούλευση σύντομα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη-μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Δεύτερη πρωτοβουλία. Η πρόταση της Κομισιόν του 2012 για την ε, ε, καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στις ε, εταιρείε που έχουν ενταχθεί, εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Μας ενδιαφέρει επίσης ιδιαίτερα η ενσχέση σας για τη διαφορά στις αμοιβέ ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών που είναι στο 16,4% αυτή τη στιγμή. Ε, πέρσι η Κομισιόν ε, ε, ε, προσπάθησε να βοηθήσει τα κράτη-μέλη στην σωστή εφαρμογή ε, των μέτρων για την μείωση αυτό, αυτής της διαφοράς στην αμοιβή και μέχρι το τέλος του χρόνου περιμένουμε να λάβουμε από τα κράτη-μέλη την την κοινοποίηση τους για τα μέτρα που έλαβαν με βάση αυτή τη σύσταση που εκδώσαμε πέρσι και μετά θα δούμε τι άλλα μέτρα θα λάβουμε. Τέλος, Χρειαζόμαστε και τους άνδρες και τις γυναίκες για να πετύχουμε τους στόχους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελο όλης της κοινωνίας. Η Κομισιόν θα εξακολουθήσει να κάνει το καθήκον της, αλλά για να πετύχουμε την ισότητα των δύο φύλων χρειαζόμαστε την προσήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των κρατών μελών καθώς επίσης και της οικονομικής του συνδρομής. Η Κομισιόν σημειώνει όλες τις συστάσεις. Θα σημειώσει όλες τις συστάσεις και θα τι λάβει υπόψη τη. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε.